Καθίστε. Καλημέρα σε όλους. Καταρχήν καλωσορίζω τον Υπουργό Μάρεκ Σαβίνσκι, προεδρεύοντα του Συμβουλίου Γεωργίας, που θα παρουσιάσει τις εργασίες και τα αποτελέσματα της Πολωνικής Προεδρίας. Αγαπητέ Μάρεκ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία σου με την Επιτροπή Γεωργίας. Συναντηθήκαμε πολλές φορές και πιο συγκεκριμένα είχαμε τρεις σημαντικές διασκέψεις, παρουσία και του Επιτρόπου Τσόλος. Συζητήσαμε όλο το νομοθετικό πακέτο το οποίο μας παρουσίασε η Κομισιόν σε αυτές τις διασκέψεις με τους υπουργούς των 27 χωρών, με τους εκπροσώπους του κλάδου και τους ακαδημαϊκούς. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και προσωπικά και εξ ονόματος της Επιτροπής για την εξαιρετική δουλειά της Πολωνικής Προεδρίας για πάρα πολλά θέματα, μερικά και πάρα πολύ δύσκολα. Πιο συγκεκριμένα να θυμίσω την πολιτική συμφωνία που καταφέραμε για το νομοθετικό πακέτο για τα γαλακτοκομικά που ήταν και το πρώτο ε, νομοθετικό ντοσιέ σε συναπόφαση το οποίο ολοκληρώσαμε. Στην επόμενη, στο επόμενο Στρασβούργο θα έχουμε την τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια και θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα. Σε ευχαριστώ Μάρεκ για την παρουσία σου και σου δίνω το λόγο για να παρουσιάσεις τα αποτελέσματα της Πολωνικής Προεδρίας. Μάρεκ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ε, βουλευτές, κυρίες και κύριοι, πέρασε ένα εξάμεινο από την πρώτη μου τοποθέτηση στην Επιτροπή Γεωργίας και τότε είχα δηλώσει ότι η Πολωνική Προεδρία θα έκανε ό,τι περνάει από το χέρι της για να προωθήσει το διάλογο μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων. Ήλπιζα σε μια καρποφόρα συνεργασία και είχα δίκιο. Ήμασταν οι πρώτη προεδρία από την οποία απαιτούσε και η συνθήκη της Λισαβόνας για πρώτη φορά στενή συνεργασία για τη συναπόφαση. Επρόκειτο για μια νέα εμπειρία και για τους ευρωβουλευτές και για τους εκπροσώπους των κρατών μελών αλλά και για την Κομισιόν. Εξαιρετικό παράδειγμα αποτελούν οι διάλογοι μεταξύ των τριών στην Επιτροπή Γεωργίας. Είχα 30 συνεδριάσεις με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την περίοδο. Κατά την Πολωνική Προεδρία είχαμε πέντε άτυπα συμβούλια γεωργίας και ε, γεωργίας για θέματα αλλίες και μετά είχαμε και ένα στο Βρόκλαβ. Και με τον πρόεδρο Ντεκάστρο συζητήσαμε τις εφαρμοστικές λεπτομέρειες που τροποποίησαν το modus operandi, τον τρόπο με τον οποίο εκτιλήσεται δηλαδή ο διάλογος μεταξύ των τριών οργάνων. Κατά την Πολωνική Προεδρία τα γεωργικά θέματα αποτέλεσαν μεγάλη προτεραιότητα με σημεία σημαντικά όπως είναι η τροφιμική ασφάλεια, η ενέργεια και η άμυνα. Εγώ προσπάθησα να ακούσω την φωνή του Ευρωκοινοβουλίου, των γεωργών, των εμπόρων στον τομέα των τροφίμων, τους καταναλωτές, και τους Υπουργούς Γεωργίας ε, της Ένωσης και των Τρίτων Χωρών. Η Γεωργία είναι πολύ σημαντική για την Πολωνία. Και οι διάφορες γνωμοδοτήσεις δεν ήταν πάντοτε ευθυγραμμισμένες ε, με τα συμφέροντά μας. Εμείς κρατήσαμε όμως την ουδετερότητά μας και λάβαμε υπόψη μας το συμφέρον της κοινότητας και ελπίζω να τα καταφέραμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την αμοιβαία συνεργασία μας στην, ε, για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Η Πολωνική Προεδρία μετά από την παρουσίαση του πακέτου από την Κομισιόν άρχισε τις εργασίες της σε όλα τα επίπεδα του Συμβουλίου, από τις άτυπες συζητήσεις μέχρι το Υπουργικό επίπεδο. Είχαμε ε, τις ε, γενικές παρουσιάσεις, τις 7 νομοθετικές προτάσεις. Τον Νοέμβριο συζητήσαμε για το νέο σύστημα των άμεσων πληρωμών και τον Δεκέμβριο συζητήσαμε για το μέλλον του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ. Και στην Ειδική Επιτροπή για τα Γεωργικά Ζητήματα κάναμε μία ανάλυση των αποτελεσμάτων της μεταρρύθμισης, δηλαδή μελέτη επιπτώσεων. Ολοκληρώσαμε και την πρώτη τεχνική ανάλυση του κανονισμού για τις άμεσες πληρωμές, την ανάπτυξη της υπαίθρου και τα χρηματοοικονομικά. Χαίρομαι που κατάφερα που κατάφερα να επεκτείνω τον διάλογο και εκτός των ορίων του Συμβουλίου διότι μπορέσαμε να συζητήσουμε από κοινού με το, Κοινοβούλιο την ε, μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ και θέλω να σας ευχαριστήσω για όλες τις ευθύνες που αναλάβατε και για την ε, καλή σας συνεργασία. Η πρώτη συζήτηση των Υπουργών με την Επιτροπή και τον, με την Επιτροπή σας και τον Επίτροπο έγινε το Νοέμβριο. Μετά έγιναν συζητήσεις με τους εκπροσώπους ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των γεωργών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Και αυτό για να μπορέσουμε να γνωριστούμε καλύτερα, να έχουμε μία αμοιβαία κατανόηση, να εμβαθύνουμε στην, στα έγγραφα σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και για το μέλλον μετά το 2013. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μία διάσταση απόψεων σχετικά με τα μεταρρυθμιστικά πακέτα για το 2013. Αυτές οι διαφορές αφορούν στην διάσταση στην, ε, στο μέγεθος της χρηματοδότησης και την κατανομή του από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα. Τα κριτήρια υποδιέρεσης ε, των ε, χρηματικών μεθόδων στον δεύτερο πυλώνα, η σύγκληση των πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντιμετώπιση των γεωργών Ορισμένες χώρες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την εναρμόνιση των πληρωμών εν ώψη του 2019. Πολλές αντιπροσωπείες ανησυχούν επίσης και για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν για τους Ευρωπαίους γεωργούς λόγω του μέτρου του greening. Ανησυχία επίσης και για τις επιπτώσεις του στην τροφιμική ασφάλεια. Επίσης θεωρούν ε, οι Γεωργοί ότι το greening ε, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικότερα ως προς τα μεγέθη του. Άλλοι ανησυχούν με το capping και αυτό λόγω των φορολογικών διαφορών στα κράτη-μέλη και των κοινωνικών διαφορών. Η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έγινε δεκτή θετικά. Ορισμένες αντιπροσωπείες θεώρησαν ότι αποτελούσαν όντως απλούστευση. Άλλες χώρες όμως είπαν ότι θα προτιμούσαν κάτι τέτοιο να είναι... Ε, να, να εναπόκειται στην διακριτική ευχή ευχέρεια του καθένα, όπως επίσης και ενισχύσεις για τους νέους γεωργούς. Η ιδέα τώρα για το τι είναι ενεργός γιοργός. Η ιδέα είναι σωστή, αλλά υπάρχουν ανησυχίες ως προς την εφαρμογή αυτού του μέτρου για να μην αυξηθεί το γραφειοκρατικό άχθος. Επίσης συζητήθηκαν τα θέματα των πληρωμών για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έθεσαν μερικοί την ανάγκη των όρων που πρέπει να τεθούν. Και ορισμένοι άσκησαν κριτικές στην Επιτροπή για την έλλειψη απλούστευσης στην ΚΑΠ. Τα μέτρα είναι πολύπλοκα, βέβαια εισάγουν νέα έναν εκδημοκρατισμό των μέτρων και διπλή προς τη θέμενη αξία. Θεωρούμε ότι η συμβολή της Πολωνικής Προεδρίας θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για τη συνέχιση του έργου αυτού από τις άλλες προεδρίες. Εμείς θελήσαμε στην Πολωνική Προεδρία να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ήπεθρο. Τον Σεπτέμβριο στο Συμβούλιο Γεωργίας η Προεδρία ξεκίνησε ένα διάλογο για την δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ε, Ευρωπαϊκής Γεωργίας εκμεταλλευόμενη την φυσικές πηγές ενέργειας. Η συζήτηση βασίστηκε ε, στα συμπεράσματα της 16ης Εβδόμου στο ΣΟΠΟΤ και στις 19 Νοεμβρίου το συζήτησαν οι Υπουργοί. Οι Υπουργοί θεώρησαν ευνοϊκά την πρωτοβουλία της Πολωνικής Προεδρίας, κυρίως την πρόταση που αφορά στην αξιοποίηση της βιομάζας. Θεωρούμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε στους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε επίσης ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να συνεχίσει να παράγει τρόφιμα. Πρέπει όμως να δούμε τι γίνεται με τα υποπροϊόντα και με τα πλεονάσματα. Είπαμε ότι έστω και αν δεν είναι δικαιολογημένο από οικολογικής ή οικονομικής πλευράς οι βιομάζες είναι σημαντική πρώτη ύλη και μπορούν να εισάγονται και από τρίτες χώρες αλλά σεβόμενες τα ίδια κριτήρια της βιομάζας που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι όλα, όλη αυτή η δουλειά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ήπεθρο θα μπορέσουν να αποδώσουν ε, ε, στη συνέχεια με τις άλλες προεδρίες. Τώρα, Πρόεδρε, σύντομα θα ήθελα να παρουσιάσω και τα αποτελέσματα των εργασιών της Πολωνικής Προεδρίας γύρω από την Πράσινη Βίβλο. Τον Ιούλιο του 2011 η Προεδρία παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο για την πολιτική πρόθεση και υποστήριξη. Για την Πολωνική Προεδρία ήταν πολύ σημαντικό ε, το θέμα της πρόθεσης ε, ευρωπαϊκών ε, γεωργικών προϊόντων στην αγορά της Ένωσης αλλά και εκτός της Ένωσης για να εγγυθούμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων. Επίσης προχωρήσαμε σε δημόσιες διαβουλεύσεις στις 29 Νοεμβρίου στην Βαρσοβία είχαμε και την τελική διάσκεψη με τίτλο «Προώθηση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας Νέα Προσέγγιση» και οργανώθηκε από την Προεδρία με την υποστήριξη της Κομισιόν. Η διάσκεψη εντάχθηκε στο πλαίσιο εργασιών της Κομισιόν για τις νέες διατάξεις που ισχύουν για την πρόθεση και πληροφόρηση γύρω από τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Στις 15-16 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο ε, αποφάσισε με τα συμπεράσματά του σχετικά με τη συνέχεια. Η συνεργασία μεταξύ των δύο των δύο οργάνων ήταν πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 2012-2013 για τους άπορους. Και αντιμετωπίσαμε δυσκολίες να βρούμε συμβιβασμό σε αυτόν τον τομέα. Είχαμε έναν άτυπο τρίλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο υποστήριξαν το συμβιβαστικό κείμενο της Πολωνικής Προεδρίας. Στις 15 Δεκεμβρίου κατά το Συμβούλιο Υπουργών καταφέραμε μετά από 3,5 χρόνια να καταφέρουμε να βρούμε μια συμφωνία σχετικά με το συμβιβαστικό κείμενο. Στο πρόγραμμα αυτό, στα πλαίσια της ΠΑΚ για το 2012-2013 Δηλαδή να μπορούμε να παρεμβαίνουμε στην αγορά και να αγοράζουμε τρόφιμα 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και να φροντίζουμε τις ε, τράπεζες ε, τροφίμων. Τώρα πάμε στο κεφάλαιο γάλα. Πριν από έξι μήνες είχα διασφαλίσει ότι η Πολωνική Προεδρία θα πάλευε για να βρεθεί ένα συμβιβασμό γύρω από το πακέτο ποιότητας. Για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων η Πολωνική Προεδρία επεξεργάστηκε ένα κοινό κείμενο με το Κοινοβούλιο με τα βασικά στοιχεία που ενισχύουν αλλά και εξαλαφρώνουν το σύστημα των σημάτων γεωγραφικής προέλευσης. Καταφέραμε να συμφωνήσουμε στον επανο, επανορισμό και στον καθορισμό του συστήματος τον ντοπ και τον ΔΟΚ. Επίσης, δώσαμε και τον, τη σήμανση ορεινό προϊόν. Επίσης, ε, ε, είδαμε ξανά τις ποσότητες των προϊόντων που πρέπει να προστατευτούν και το θέμα, είπαμε, της γεωγραφικής προέλευσης. Η Πολωνική Προεδρία εξετάζει προσεκτικά τις θέσεις που έχουν υποβληθεί αλλά οι αποφάσεις ε, θα ληφθούν σύντομα από την Δανέζικη Προεδρία. Καταφέραμε όμως επί Πολωνικής Προεδρίας να βρούμε μία μίνιμουμ συμφωνία. Εκρεμεί όμως ε, το θέμα της ε, γεωγραφικής προέλευσης που πρέπει να αποτελέσει ένα εμπορικό στοιχείο πλέον και το έχει στα χέρια της το θέμα η Δανέζικη Προεδρία. Η Πολωνική Προεδρία και η Κομισιόν κατάφεραν να βρουν συμφωνία και για το γάλα στον τρίλογο της 6 Δεκεμβρίου του 2011. Εξάλλου εσείς μιλήσατε γι' αυτό. Και στο τέλος για την μερικά λόγια για την προσαρμογή των γεωργικών διατάξεων στη Συνθήκη της Λισαβόνας το Ξάμιν αυτό η Πολωνική Προεδρία προσπάθησε να καταλήξει σε συμφωνίες, οριζόντιες συμφωνίες για την προσαρμογή με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είχαμε διάφορες συνεδριάσεις σχετικά και πιστεύουμε ότι καταφέραμε να επεξεργαστούμε έναν ορίζοντα για την οριζόντια εφαρμογή τεσσάρων βασικών διατάξεων της ΚΑΠ. Είχαμε στα τέλη Δεκεμβρίου έναν τελευταίο τρίλογο και μου φαίνεται ότι πλέον η συμφωνία είναι στην πόρτα. Λοιπόν, ας φτύσουμε στον κόρφο μας και ας ελπίσουμε ότι επί η Προεδρία θα λυθεί το πρόβλημα. Για να μπορέσουμε δηλαδή να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να προχωρήσουμε και στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ λύνοντας όλες τις εκκρεμότητες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία εκκρεμούν, τα οποία δεν θα τα αναφέρω εδώ σήμερα. Στόχος μας κατά την Προεδρία ήταν να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προκλήσεις ως Προεδρία. Ελπίζω ότι συνεισφέραμε συνεισφέραμε και στις γευστικές σας ε, στις, και προκαλέσαμε και τη γεύση σας μάλλον καλύτερα αυτό το εξάμεινο προσπαθώντας να σας γνωρίσουμε όταν μιλούσαμε για τη γεωγραφική προέλευση όλα αυτά τα καλά πολωνικά προϊόντα όπως οι φράουλες της Κασούμπα. Ελπίζω ότι δώσαμε ένα καλό έναυσμα στη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Εγώ δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Πρόεδρε αλλά και όλους τους βουλευτές αυτό το εξάμεινο ελπίζω μάλλον ότι η γραβάτα που προτείνουν οι Δανείοι ως σουβενίρ της προεδρίας τους να είναι μια γραβάτα ευίωνη και να μπορέσει να σας βοηθήσει να λύσετε όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και ευχαριστώ και για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες σχετικά με τις συζητήσεις που έγιναν στο Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, για τις κριτικές, για τις δυσκολίες, πράγματα τα οποία θα θησαυρίσουν όλοι μας οι εισηγητές για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν Στη συνέχεια εσύ θέλησες να υποστηρίξεις ένα διάλογο ως Πολωνική Προεδρία και σε ευγνωμονούμε πρόκειται για μια νέα εμπειρία αυτή της Λισαβόνας και για το Κοινοβούλιο, όχι μόνο για το Συμβούλιο. Είναι καλό λοιπόν ε, να ξέρει ο καθένας ε, να, τις θέσεις ε, του άλλου για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις γρήγορες αλλαγές που χρειάζεται ο γεωργικός κόσμος της Ευρώπης. Το πακέτο γάλαγα αποδεικνύει ότι η συναπόφαση δεν παρέτεινε τους χρόνους έγκρισης των προτάσεων. Δεκέμβριος 2010 η πρόταση της Κομισιόν 6 Δεκεμβρίου 2011 η τελική συμφωνία. Μέσα σε ένα χρόνο εγκρίναμε ένα νομοθετικό κείμενο και αυτό λόγω της ε, καρποφόρα συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ξεκινάμε τη συζήτηση, έχουν γραφτεί πολλοί συνάδελφοι. Ο Άλμπερ Ντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα για να μας παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της Πολωνικής Προεδρίας που εντυπωσιακά. Μας είπατε ότι η Πολωνία για πρώτη φορά κατήχε την Προεδρία. Να σας πω ότι ήταν καλή η Προεδρία. Οι τριμερείς διάλογοι στους οποίους αναφερθήκατε δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Οι πολλαπλές συναντήσεις με το Κοινοβούλιο στο πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας, καταρχάς μεταξύ της Επιτροπής ε, ε, Γεωργίας και των Υπουργών Γεωργίας. Σημείωσα και αυτά που είπατε, ότι και το δικό σας ε, έργο το διακατήχε πνεύμα κοινοτικό. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν αυτό τον κοινό ευρωπαϊκό στόχο να ακολουθήσουμε για να υπάρχει μέλλον στην ε, κοινή γεωργική πολιτική και σε αυτό θα σας υποβοηθήσουμε. Πολλά από αυτά που είπατε τα υποστηρίζω απόλυτα. Συμφωνώ και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των σημερινών προτάσεων. Εδώ, ως Κοινοβούλιο και ως Συμβούλιο, πολλά έχουμε να κάνουμε προκειμένου η μεταρρύθμιση να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο να μην ε, προκύψει πιο πολύ γραφειοκρατία, αλλά πιο λίγη γραφειοκρατία. Σας εύχομαι και στη συνέχεια κάθε επιτυχία στο έργο σας για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και ελπίζω μετά το τέλος της Πολωνικής Προεδρίας να διατηρήσετε τις επαφές με την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου από κοινού Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να συνεργαστούμε για το μέλλον της ε, αγροτικής πολιτικής. Σας εύχομαι και σε προσωπικό επίπεδο κάθε επιτυχία γιατί ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία η συνεργασία μαζί σας και ελπίζω να συνεχίσουν οι επαφές σας. Ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. E ε, ευχαριστώ Ο Λουίς Κάπουλα Σάντος. <coughs> e do meu grupo político, Και προσωπικά και εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους, τους Πολωνούς, για την προεδρία τους. Προσωπικά μπορώ να πω ότι το στοιχείο διαφοροποίησης των πολιτικών που ασχολούνται με τη γεωργία και την Ήπεθρο είναι το πάθος. Μπορούμε λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι ο Υπουργός ο Πολωνός συμμερίζεται το πάθος που έχουμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη γεωργία. Μπορώ λοιπόν τώρα να συγχαρώ τους Πολωνούς για την εμπειρογνωμοσύνη την οποία επέδειξαν και την τεχνική τους επάρκεια. Η Πολωνική Προεδρία έκανε ό,τι μπορούσε και για να κλείσει ορισμένα κεφάλαια και για να ξεκινήσει τη συζήτηση σε ορισμένα θέματα. συμμερίστηκαν οι Πολωνοί και με κάποιες ανησυχίες που έχω εγώ όπως η μικρή λεγόμενη γεωργία, ο αγροτουρισμός κτλ. Ο απολογισμός των Πολωνών λοιπόν είναι θετικός. Ήταν μια έκπληξη συνολικά θετική, μπορώ να πω, η Πολωνική Προεδρία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια των δραστηριοτήτων σας Κύριε Υπουργέ, εύχομαι ότι η μαχητικότητά σας και η ενέργειά σας θα συνεχίσει να είναι χρήσιμη και θα μπορέσουμε έτσι να ωφελήσουμε την Ευρωπαϊκή Γεωργία και την Ήπεθρο της Ευρώπης. Έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και μια ουσιαστική, θα έλεγα, συμμαχία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι και οι επερχόμενες προεδρίες θα αναγνωρίσουν στην Γεωργία την σημασία που επεδείξατε εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους Πολωνούς όπως και οι προηγούμενοι προλαλήσαντες Νομίζω ότι όλοι εξεπλάγημεν θετικά από το ποσοστό εμπλοκής το οποίο εσείς προσωπικά επιδείξατε και τη συνεργασία σας με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας. Σας συναντήσαμε επανειλημμένα, είχαμε πολύ σοβαρές συζητήσεις μαζί σας. Συζητήσαμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις της για την μεταρρυθμίσεις στην ΚΑΠ. Δείξατε προθυμία στην επαφή μαζί μας και είχατε και υψηλά θα έλεγα επίπεδα ολοκλήρωσης των φακέλων με τα οποία ασχοληθήκατε. Νομίζω ότι αυτά που κάνατε εσείς είναι ένας πρόδρομος θα έλεγα και σε σχέση με τα CMO. Είναι ένα πρώτο βήμα για το τι θα ακολουθήσει έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις κρίσεις των αγορών που άρχισαν να εμφανίζονται τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Με λίγα λόγια, το κλίμα συνεργασίας ήταν εξαιρετικό. Δεν θα σας χάσουμε τους επόμενους μήνες, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα μαζί και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια νέα ΚΑΠ η οποία θα είναι μάρτυρας μιας ευημερούσας Ευρώπης. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Χοισλέν, θα ήθελα να σας χαρώ για την Προεδρία σας, να συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Ε, θέσατε ένα, αν θέλετε, πρότυπο για τις συζητήσεις ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ήταν πραγματικά κάτι εντελώς καινούριο αυτή, η συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής μας και των Υπουργών Γεωργίας και καταλάβαμε τουλάχιστον ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον το Κοινοβούλιο. Οι συζητήσει ήταν τόσο καρποφόρες ε, και καταλαβαίνουμε τις ε, θέσεις σας, τις καταλάβαμε πολύ καλύτερα. Ελπίζω ότι και εσείς τα καταλάβατε καλύτερα κάποιες πράσινες θέσεις προκειμένου αυτή η διαδικασία του διαλόγου να συνεχιστεί, ελπίζουμε. Νομίζω ότι μετά από την υποβολή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, γεωργική πολιτική, βασικά προβλήθηκε η κριτική. Οι επικριτές ε, ακούγονται πολλοί, αλλά εμείς ελπίζουμε να ακουστούν και αντιπροτάσεις, να κατατεθούν εναλλακτικέ ε, προτάσεις. Γιατί αν δεν το κάνουν αυτό άλλοι, θα πρέπει ε, το Κοινοβούλιο να καταθέσει θετικές εναλλακτικέ προτάσεις. Ε, Για αυτό το σκοπό συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα του πακέτου ποιότητα. Δυστυχώ δεν προχωρήσαμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο της ε, πολιτικής και στα θέματα και ετικετοθεσίας να προχωρήσαμε, δυστυχώς. Ήταν διαφορετική στάση που επικράτησε στο Συμβούλιο. Γνωρίζω τα προβλήματα που επικρατούν και στην ίδια μου τη χώρα. Σε άλλα πακέτα, για το γάλα για παράδειγμα, δεν μπόρεσε να συμφωνήσει η ομάδα μας ε, δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, αν θέλετε, για το γάλα. Διαφαίνεται στον ορίζοντα και η επόμενη κρίση, άλλωστε, για θέματα γάλακτος. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια ρύθμιση της αγοράς στον κλάδο αυτό. Σας εύχομαι λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η ανοιχτή συνεργασία η οποία διέπεται από εμπιστοσύνη ακόμα και αν δεν θα ηγείστε πλέον αλλά να ξέρετε ότι οι βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι στη διάθεση της Πολωνίας για συζήτηση για θέματα αγροτικά γιατί είναι πολύ σημαντική γεωργική χώρα η Πολωνία χωρίς την Πολωνία δεν θα μπορέσει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση και ελπίζουμε να έχουμε την υποστήριξή σας στο πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστώ εκ νέου για την πολύ καλή συνεργασία. Grazie Martin, è arrivato Jim. Jim Nicholson alla parola. Ο Jim Nicholson έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον Υπουργό γιατί ως εισηγητής το πακέτο για τα γαλακτοκομικά εξαρτώμουν ιδιαίτερα από το προσωπικό της Πολωνικής Προεδρίας και του Συμβουλίου. Θα ήθελα πραγματικά να τους επενέσω για τον τρόπο με τον οποίο ολοκλήρωσαν και διεξήγαν τα καθήκοντά τους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο αυτό σε εποχές που ήταν πάρα πολλέ πολύ ενδιαφέρουσε να το θέσω έτσι. Αλλά οι υπάλληλοι σα πάντα μας ε, βοήθησαν. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία στην Προεδρία σας. Θα υπογραφεί ίσως την άλλη εβδομάδα και έτσι δεν θα δράξετε ένα μέρος της δόξας που θα σας άρμοζε, αλλά θα σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για τη συνεργασία. Νομίζω ότι για όλες τις πλευρές η περίοδος αυτή και το θέμα αυτό μας δίταξε πολλά. Ήταν ίσως το πιο μεγάλο θέμα υπό συναπόφαση. Στην αρχή δεν ήμασταν όλοι βέβαιοι για το πώς, αντιδράσει, πώς θα αντιδράσει η άλλη πλευρά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το έργο αυτό, δυσκολευτήκαμε πολύ, αλλά σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά άλλα συμβαίνουν παράλληλα στην Ευρώπη ασφαλώς και ασφαλώς έχουμε φτάσει μέσα Ιανουαρίου και θα πρέπει να παραδεχτώ ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώνεται η κατάσταση ως διαμορφώνεται σε θέματα αγροτικά θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί και είναι αξιοθαύμαστο ότι έχουμε δύο μέλη από τον Εμένο Βασίλειο στην κυβέρνηση που ήταν εδώ στο Κοινοβούλιο όταν εγκρίθηκε η νομοθεσία. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι επικρατούν ίδιες συνθήκες για όλη την κτηνοτροφική βιομηχανία σε ό,τι αφορά τους κλωβούς στοιχείων, τις στοιχείες κλωβών. Μιλάμε για θέματα ευημερίας των ζώων, πολύ βασικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα ο λόγος στον κύριο Ανιώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε ο Τζιμ Νίκολσον. Ευχαριστούμε τους Πολωνούς και τον Υπουργό Γεωργίας. Θέλουμε πραγματικά όμως να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό. Σχετικά με την κατανομή των άμεσων πληρωμών τώρα, προέρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαδικασία εξο... αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθεί. Αν ήμουν ο Υπουργός Γεωργός, ο Υπουργός ε, της Γεωργίας της Πολωνίας, οι δυσκολίες που θα είχα να αντιμετωπίσω ε, ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Σας είχαν υποσχεθεί ότι θα υπήρχε η διαδικασία αυτή εξίσωσης και σε εσά και στους Λιθουανούς, Λετονούς κτλ. Αλλά στην ουσία δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Αυτό αποδυνάμωσε την πίστη την οποία έχετε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο ασκήσατε την Προεδρία σας. Δείξατε σε αυτούς οι οποίοι αμφέβαλαν την πίστη που τρέφει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η μεγάλη χώρα σας. Είχα την τιμή να συμμετέχω στην ομάδα που διαπραγματεύτηκε μαζί σας το πακέτο γαλακτοκομικών. Μάθαμε πολλά και τα μάθαμε μαζί θα έλεγα. Ήταν μια διαδικασία μαθητείας σε επίπεδο συναπόφασης. Η ερώτησή μου λοιπόν αφορά περισσότερο τη μέθοδο εργασίας. Όπως είπα έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία μαθητείας και εσείς και οι συνεργάτες σας κάνατε ό,τι μπορούσατε, δείξατε πολλή ενέργεια για να καταφέρετε να καταλήξετε σε κάποιες συνενετικές προτάσεις στο Συμβούλιο. Μια από τις δικές μας δυσκολίες στο Κοινοβούλιο ήταν ότι το Συμβούλιο δεν σας έβαζε σε καλή θέση διαπραγμάτευσης λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα είναι δυνατόν να βελτιωθούν οι συνθήκες συνεργασίας για να έχουμε μια συναπόφαση ταχυτέρα και αποτελεσματικότερη. Σίγουρα αυτό που ζήσαμε μαζί δεν ήταν ταχύ μεν, αλλά ήταν αρκετά αποτελεσματικό. Ο κύριος Γιάρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρα, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον ε, Πολωνό Υπουργό. Θα ήθελα να τονίσω, πέρα από αυτά που ακούσαμε, ότι η δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου με το Κοινοβούλιο πραγματικά έθεσε πρότυπα, πραγματικά καταφέραμε να συζητήσουμε. Έτσι λοιπόν φανταζόμαστε τη δημοκρατία, έτσι φανταζόμαστε την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Γι' αυτό λοιπόν και ευχαριστώ την Προεδρία σας. Μία έκκληση, μία παράκληση. Με μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσα ότι ε, μας παρουσιάσατε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΚΑΠ και μας είπατε ότι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα στην εφαρμογή, κυρίως ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν σας απευθύνω την εξής έκκληση. Αφήνετε τα ενία της Προεδρίας, αλλά συνεχίζετε να συμμετέχετε με την εμπειρία σας. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ μην αμελήσετε ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν και θα πρέπει να τα υποστηρίξει και η διοίκηση αλλά και τελικά οι αγρότες μας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια βιώσιμη υποστήριξη. Μην αμελήσετε λοιπόν το θέμα αυτό της εφαρμογή και πάλι σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βλάσοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αίσθησή μου είναι ότι μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε για την Προεδρία, μετά από όλα τα σχόλια των συναδέλφων, μπορείτε να είστε ικανοποιημένοι. Βέβαια δεν απευθύνονταν μόνο σε εσά, γιατί και όλοι οι τεχνικοί οι οποίοι σας συνόδευαν και όλοι οι διπλωμάτες και αυτοί ε, ε, πρέπει να τύχουν συγχαρητηρίων. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω ένα ερώτημα τώρα. Στις 4 Σεπτεμβρίου στην Τσεστόχοβα, στην Πολωνία, σε μια ομιλία σας είχατε πει ότι θα αναλυφθεί δράσεις έτσι ώστε η Ευρώπη να απαλλαγεί από γενετικά τροποποιημένα. Τι μέτρα πήρατε σαν Προεδρία για να εφαρμόσετε τη συγκεκριμένη σας ρίση. Ευχαριστώ κύριε Βλάσοβιτς, αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Δίνω και πάλι το λόγο στον Μάρεκ Σαβίνσκι για να απαντήσει. Και επαναλαμβάνω τα συγχαρητήριά μου και τους επένους μου για την εξαιρετική δουλειά. Ο Μάρεκ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, Ευχαριστώ για όλες τις τοποθετήσεις. Ευχαριστώ και για τους επένους και για τις πιο επιφυλακτικές τοποθετήσεις. τα, τα αιτήματα των δύο Βρετανών βουλευτών για την ευημερία των ε, πουλερικών σε κλωβοστοιχίες ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως για την Πολωνία, διότι μας δαχτυλόδεχναν εδώ και καιρό. Αλλά εμείς εξυγχρονίζουμε τα ορνηθοτροφία μας ε, στην Πολωνία. Δεν θα τα καταφέρουμε βέβαια μέχρι, δεν τα καταφέραμε μέχρι το τέλος του 2011. Αλλά μέσα από μία συμφωνία κυρίων είπαμε ότι μέχρι το 2012 θα τα έχουμε καταφέρει. Στην Μεγάλη Βρετανία... Ήσασταν οι πρωτοπόροι στην τροποποίηση του συστήματος εκτροφής των ορνήθων. Τώρα, μετά από την πενταετή μου εμπειρία στο Συμβούλιο και το εξάμεινο της Πολωνικής Προεδρίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αναζήρω το τελευταίο μου συμπέρασμα. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο για μια τεράστια συζήτηση. Και ας μην τα βάζουν μαζί μου οι υπάλληλοι, αλλά πολλές φορές οι προτάσεις που υποβάλλουν και μας τις παρουσιάζουν έτοιμες, είναι ένα copy-paste, ένα κόψε και κόλλα ε, παλαιών προτάσεων. Το, μη με παρεξηγείτε γι' αυτό, αλλά το θέμα της ευημερίας των ζώων, όπως και η μεταρρύθμιση της χρειάζονται άτυπες συνεδριάσεις όπου δεν μας περιορίζεται ο χρόνος, όπου δεν έχουμε δύο ή τρία λεπτά για κουβέντα. Όχι, χρειάζεται ανοιχτή συζήτηση με επιχειρηματολογία, ο καθένας να παρουσιάζει τους λόγους του. Εχθές με το έναυσμα της Δανέζικης Προεδρίας, με μία σύντομη συνεδρίαση σε ένα πρωινό μπροστά σε ένα μπουφέ, Ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών με ρώτησε να τον ενημερώσω για το πώς έχουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Και μου είπανε, μα με 500 εκατομμύρια κατοίκους δεν το φαντάζεστε καν ότι θα έπρεπε να έχετε τουλάχιστον ένα πόθεμα σταριού. Δεν κρατάτε, δεν τηρείτε εσείς οι ήδη τις αρχές που επιβάλλετε σε τρίτες χώρες. Μπορείτε εσείς να εξαρτάστε έτσι από τρίτες χώρες για τέτοια θεμελιώδη είδη διατροφής και δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι που μας τα ρωτάνε και εμείς ίδιοι αναρωτιόμαστε πολλές φορές τι γίνεται. Οι γεωργοί μας, ας πούμε, να, οι Πολωνοί γεωργοί του αναρωτιούνται. Δηλαδή ένας γεωργός έχει τη γεωργική του εκμετάλλευση για να παράγει. Και από 15 χρόνια η βασική πηγή των εσόδων του ήταν η παραγωγή του. Σήμερα το βασικό εισόδημα των γεωργών προέρχεται από τις άμεσες πληρωμές. και προηγείται και το θέμα της εναρμόνισης. Ναι, οι Πολωνοί, οι Γεωργοί μιλάνε για το επίπεδο των πληρωμών. Και τους έλεγα εγώ, κοιτάστε, εκπροσωπώ όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό το οποίο λέω εγώ σήμερα είναι μήπως τελικά όλο αυτό το σύστημα πληρωμών είναι αυτό το οποίο διαταράσσει συνολικά όλο το ανταγωνιστικό κεφάλαιο. Δεν θα έπρεπε ίσως να μείβονται οι δραστηριότητες, να γίνονται ή πληρωμαίες με διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, 7% αγρανάπευση. Η πληρωμές με διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, 7% αγρανάπαυση. Η αγρανάπαυση πρέπει να είναι υποχρεωτική Δεν θα έπρεπε τα κονδύλια να πάνε προς αυτό το 30% των γιοργών οι οποίοι θέλουν να εισάγουν στις εκμεταλλεύσεις του καλλιέργειες ε, ε, ε, πρωτεϊνούχων φυτών Δηλαδή, ας σταθούμε λίγο σε, αυτές, σε αυτά τα στοιχεία υποχρέωσης και ελεύθερης επιλογής. Όλη αυτή η προβληματική θα ξανάρθει επιτάπητος, διότι είναι ασύλληπτο να λέμε ότι νύπτουμε τα χείρα μας διότι κάθε χώρα πρέπει να αποφασίζει μονάχη της. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο σήμερα διότι η αγορά είναι παγκόσμια. οι γενονετικά τροποποιημένοι οργανισμοί λένε ότι καταστρέφουν τη βιοπικιλότητα και μπορεί να είναι επιβλαβής ε, για την υγεία. Γιατί η Ευρώπη φοβάται να καλλιεργεί γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς για να μην πειράξει τη δικιά της βιοπικιλότητα ενώ ανέχεται την καταστροφή της βιοπικιλότητας των άλλων και εισάγει ζωοτροφές από αυτές τις τρίτες χώρες εγώ πολλές φορές το συζήτησα αυτό με τους συναδέλφους υπουργούς και ελπίζω ότι θα υπάρξει συζήτηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Κύριοι βουλευτές, το εξάμεινο που πέρασε αποτέλεσε πολύ σημαντική προσωπική εμπειρία και για μένα αλλά και για σας και όχι μόνο τους Πολωνούς Ευρωβουλευτές και για τους υπαλλήλους η κεκτημένη εμπειρία ελπίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί σωστά και υπέρ όλων στη συνέχεια των εργασιών μας για μια Ευρώπη πιο ωραία και πιο σύγχρονη. Ευχαριστώ Μάρεξ, ευχαριστώ για τη συζήτηση, ευχαριστώ και τους συναδέλφους που μίλησαν. Ήταν μια πολύ θετική εμπειρία και ευχόμαστε η Δανέζικοι Προεδρία να αναπάρει τη σκητάλη από την Πολωνική Προεδρία και να συνεχίσει κατά τον ίδιο τρόπο τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Διακόπτουμε για, για μερικά λεπτά, ούτω ώστε να φύγει ο κύριος Σαβίνσκι και μετά θα συνεχίσουμε με το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη. Ο Σπύρος Δανέλης είναι εδώ. Λίγα λεπτά μόνο. Allora riprendiamo i lavori. Bene, possiamo riprendere i lavori. Punto 8 all... Ευχαριστώ. Σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη. Το εμπόριο για την αλλαγή επενδυτική στρατηγική για τον Μεσογειακό Νότο μετά την Αραβική Άνοιξη, μετά, τη... ναι, μετά την Αραβική Άνοιξη, ο Σπύρος Δανέλης. Πάμε λοιπόν για, στην εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Μεσογειακό Νότο μετά την Αραβική Άνοιξη. Κατά την τελευταία συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου η συζήτηση για αυτό το σημείο αναβλήθηκε για τεχνικούς λόγους. Όπως όλοι γνωρίζετε, το σχέδιο αλλαγής ε, της, ε, του Μεσογειακού Νότου μετά την Αραβική Άνοιξη είχε σημαντικές επιπτώσεις και για την Ευρωπαϊκή Άνοιξη Χρειάζεται λοιπόν ε, η φορεία και ανάπτυξη στην περιοχή για να εγγυθούμε δημοκρατία και πολιτική σταθερότητα. Η γεωργία και η ανάπτυξη πέθρου είναι πολύ σημαντικές σε αυτή τη διαδικασία σταθεροποίησης, διότι συμβάλλουμε στην ε, τροφιμική ασφάλεια, στην κατανομή δίκαιων εσόδων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δίνω το λόγο στο Σπύρο και ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Και μετά την τοποθέτηση του Σπύρου Δανέλη θα γίνει συζήτηση, μετά θα ακούσουμε την Κομισιόν και θα περάσουμε μετά στο τελευταίο σημείο που είναι το σημείο 9. Ο Σπύρος. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας για την επικοδομητική συνεργασία μας. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα, που όπως σωστά είπατε πρόεδρε είναι εξαιρετικά σοβαρό και σε αυτή τη συγκυρία ιδιαίτερα. Ως γνωστό η διεργασία των αλλαγών στη Νότια Μεσόγειο που ξεκίνησε με την Αραβική Άνοιξη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και είναι μάλλον αβέβαιο ε, για το αν θα οδηγήσει και πότε τελικά σε θεμελίωση της δημοκρατίας και της πολιτικής σταθερότητας που βεβαίως αποτελεί και στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη πολιτικής σταθερότητας είναι μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας και η ανάπτυξη πέθρου είναι καθοριστική στις διεργασίες σταθεροποίησης, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες αυξημένης αστάθειας στις παγκόσμιες αγορές. Και αυτό διότι η ανάπτυξη αυτών των τομέων βοηθά στην προώθηση της επισητιστικής ασφάλειας, σε μια πιο δίκαιη δημιουργία και κατανομή του εισοδήματος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ένταξη των γυναικών και των μικροκαλλιεργητών στην οικονομία, που συνιστά βεβαίως ένα κρίσιμο παράγοντα για τη δημιουργία και διάχυση εισοδήματος σε αυτό το στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλώς θα πρέπει να βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να βρει και τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επιτευχθεί αύξηση του εισοδήματος και η διάχυσή του στην περιοχή, ώστε να επιτευχθεί καταρχάς ο στόχος της επισητιστικής ασφάλειας. Βεβαίως δεν αρκεί να υπάρχει τροφή. Πρέπει να υπάρχουν και τα χρήματα για να την εξασφαλίσουν. Όπως και με την τεχνογνωσία, ισχύει ότι δεν αρκεί η παραγωγή της, αλλά απαιτείται και η ευρεία διάχυση της γνώσης, ώστε αυτή να φέρνει και αποτέλεσμα. Απαιτείται λοιπόν όχι απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την πρόθεση επενδύσεων στον τομέα των υποδομών, παραδείγματος χάρη αρδευτικά έργα, υποδομή για επεξεργασία, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορά προϊόντων και συστήματα εμπορίας, η μεταφορά της γνώσης και βελτιώσεις τους θεσμούς. Και θα πρέπει βέβαια σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να αποφευθούν εύκολες και βραχυπρόθεσμες λύσεις που θα έδιναν αποτελέσματα μη συμβατά με τη διεθνή επιδίωξη για βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και της ενέργειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Μια τέτοια στρατηγική δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει την ανάπτυξη του εμπορίου προς αμοιβαίο όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής της Νότιας Μεσογείου. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό αυτή η ανάπτυξη να προωθείται όχι μόνο εξασφαλίζοντας προνομιακή πρόσβαση σε περισσότερα προϊόντα, αλλά και σε βάθος, εξασφαλίζοντας δηλαδή σύγκληση στα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Μεσογείου κανονιστικά πλαίσια σχετικά με την παραγωγή, το εμπόριο αλλά και άλλους τομείς της οικονομίας. Και βέβαια θα πρέπει μια τέτοια ανάπτυξη να λαμβάνει υπόψη τις, συνέπειες στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στους ευαίσθητους τομείς της. Τέλος, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεσολαβήσει ώστε να αποφευχθούν μονομερείς κινήσεις που επηρεάζουν το εμπόριο και αποσταθεροποιούν τις διεθνείς αγορές, καθώς και για να αναπτυχθεί ένα περιφερειακό μοντέλο ανάπτυξης του εμπορίου μεταξύ των χωρών της Βορείου Αφρικής και των χωρών νοτίως της Σαχάρας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο. Σε ευχαριστώ για την παρουσίασή σου. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Η Γέγκερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή, τον κύριο Δανέλη, για αυτά τα οποία μας είπε, για τις εξηγήσεις του δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει γιατί τα θέματα αυτά πρέπει να συζητηθούν στην Επιτροπή μας. Στη φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα ξέρετε ότι συζητάμε και θα περάσουμε στην αρμόδια Επιτροπή στην ψηφοφορία της εμπορικής σχέσης, τη σύναψη μάλλον και ε, της εμπορικής συμφωνίας με το Μαρόκο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συγκεκριμένη χώρα και φυσικά για μας το εμπόριο παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο φυσικά στις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές. Βέβαια δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για το εμπόριο, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την εμπορική δραστηριότητα. Υπάρχει το θέμα των ανθρώπων, υπάρχει το θέμα των πολιτών, υπάρχει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία ε, ε, προασπίζει η Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μιλάμε για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κρατος δικαίου, δημοκρατία και όλα αυτά. Είπατε και μιλήσατε για την δική κατανομή των εισοδημάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Τι σημαίνει ότι η παραγωγή, δηλαδή οι μικροί αγρότες, θα είχαν πιο πολλές ευκαιρίες, δυνατότητες. Αυτό ως τώρα πραγματικά δεν αρκεί, πολύ απλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να υπάρχει πραγματική πρόσβαση στις, ε, στους πόρους, στις ποσοστώσεις. Μιλήσατε για ε, μια σύγχρονη μορφή υδροδότησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει στον τομέα αυτό να ζητήσουμε και οικολογική ανάπτυξη. Ακόμη και στη γεωργία. Ιδάλλως θα υπάρξουν και άλλες λύσεις ενδεχομένως με τις οποίες σκέφτομαι και την ενέργεια θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τον κλάδο και να μας υποστηρίξουν και άλλοι κλάδοι. Θα ήθελα να ευαισθητοποιήσω με τη σύμβολή μου να μην κοιτάξουμε μόνο το εμπόριο και τα χρήματα πάντα να έχουμε υπόψη μας τι κάνουν οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από τις συμφωνίες αυτές και πίσω από τις εκθέσεις αυτές τις οποίες συζητάμε. Και θεωρώ ότι ακόμα και στην ομάδα μου δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη για τα στοιχεία αυτά. Δεν μπορούμε μόνο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να μιλάμε για εκδημοκρατισμό, για κρατικό δικαίου. Όχι. Θα πρέπει αυτό να εφαρμόζεται εγκάρσια σε όλες τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα ήθελα να υπερασπίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους υπόλοιπους συναδέλφους, εφόσον θέλουν το λόγο, ο κύριος Μποβέ. Ναι, ήθελα να ζητήσω το λόγο σχετικά με την έκθεση <clears throat> του κύριου Δανέλη και ίσως να προσπαθήσω να φωτίσω λίγο περισσότερο αυτά τα οποία ακούστηκαν τους προηγούμενους συναδέλφους. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Εάν πράγματι θέλουμε να στηρίξουμε τις χώρες αυτές είναι για να τις βοηθήσουμε, τις χώρες του Μαγκρέμπ και του Μασρέκ, να προχωρήσουν και να κάνουν πρόοδο στον τομέα της ασφάλειάς τους στην προμήθεια τροφίμων. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να οργανωθούν περιφερειακά, σε μια περιφερειακή αγορά. Το θέμα των περιφερειακών αγορών είναι θεμελιώδες. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές της Μεσογείου με στόχο την τροφιμική επάρκεια. Πρέπει να υπάρξουν περιφερειακές συμφωνίες ανάμεσα στις χώρες αυτές και την υποσαχαρική Αφρική ίσως. Θα δούμε. Νομίζω ότι το θέμα των δικαιωμάτων επίσης είναι κάτι το θεμελιώδες. Μιλάμε για την πρόσβαση στην γη, την καλλιεργήσιμη γη, αυτό είναι προτεραιότητα. Ο κίνδυνος είναι κάποιες από τις κυβερνήσεις που δεν έχουν χρήματα, είναι έτοιμες να εκχωρήσουν τεράστιες γέες. Είδαμε τι έγινε στο Μαρόκο δυστυχώς, βλέπουμε ότι θα γίνει και σε άλλες χώρες και αυτό μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια σε τρόφιμα. Πρέπει λοιπόν να διασφαλιστεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς. Τώρα, ο σεβασμός των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι σε πολλές από τις χώρες αυτές δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδιαίτερα των ημερομίσθιων εργαζομένων και των ε, διαδικασιών επεξεργασίας τροφίμων κτλ. Τώρα για τους υδάτινους πόρους. Ξέρετε ότι γενικά μιλάμε για εκμετάλλευση υδάτινων πόρων σε πολύ μεγάλο βάθος, χωρίς αντικατάσταση των πόρων αυτών. Και γι' αυτό αν υπάρχει εντατική και απρόβλεπτη χρήση των πόρων αυτών δεν θα υπάρξει ανανέωσή τους. Στην Ευρώπη λοιπόν έχουμε αναπτύξει κάποια καινοτόμα προγράμματα χάρη στο πρόγραμμα LEADER στα leader λοιπόν, εγώ θα ήθελα στα πλαίσια της πρότασης που κάνουμε να χρηματοδοτήσουμε και κάποια μεσογειακά leader, ίσως και συνδεδεμένα με τα δικά μας leader, για να επιτρέψουμε την αυτοοργάνωση των παραγωγών των γεωργών, να μην τους αφήσουμε αδύναμους απέναντι στις αγορές, αλλά να βοηθήσουμε να προωθηθεί η οργάνωση των παραγωγών στις χώρες αυτές, ε, και στα εδάφη των χωρών της Νότιας Μεσογείου. Να βλέπουμε δηλαδή το θέμα όχι μόνο σαν τομής παραγωγικότητας, αλλά εδαφικά, συνολικά, σε περιφέρεια. Θα ήθελε κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Κλάρκ έχει το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ιδιαίτερα την γνωμοδότηση του κυρίου Ντανέλη. Είναι πολύ ισορροπημένη και συμφωνούμε με την απόψη που εκφράζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η σχετική ε, εμπορική στρατηγική ως προς τις επενδύσεις και μπορεί και πρέπει να επηρεάσει τις εξελίξεις στην Νότιο Μεσόγειο, σαφέστατα. Συμφωνούμε με τον κύριο Δανίλη ότι ως τμήμα της στρατηγικής αυτής και της διαδικασίας αυτής φυσικά θα πρέπει να ανοίξει περαιτέρω η αγορά και αυτό ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει την ε, βιώσιμη ανάπτυξη την, ε, τα δικαιώματα των μικρών αγροτών, τα δικαιώματα των γυναικών και του καθεξής. Αλλά πιστεύουμε επίσης, όπως ο κ. Δανέλης, ότι η πρόσβαση στην αγορά στον τομέα αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα. Η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε μεγάλο βαθμό ανοιχτή στην παραγωγή και στις εξαγωγές από την Νότια Μεσόγειο και δεν μπορούμε ασφαλώς να γνωρίσουμε και τους ευαίσθητους τομείς στο εσωτερικό της Ένωσης. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι θεωρούμε ότι το περαιτέρω άναγμα των αγορών δεν αποτελεί πανάκια. Πολύ πιο σημαντικό και αυτό σωστά το τοποθετεί η γνωμοδότηση. Πολύ πιο σημαντική είναι η επικέντρωση ε, στα μέτρα προώθηση της ανάπτυξης της υπαίθρου στις χώρες αυτές για την ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών, όπως μόλις ανέφερε ο κύριος Μποβέ, για την βελτίωση της ασφάλειας, της επιστημιστικής ασφάλειας και γενικότερα η συνεργασία με τις χώρες αυτές για την ανάπτυξη θεσμών σε ό,τι αφορά τον κλάδο της αγροτικής ανάπτυξης προκειμένου σταδιακά και βαθμία να μπορέσουν να εναρμονιστούν με το κινητικό και εκτιμένο και την ε, κοινή ακροτική πολιτική. Επ' αυτόν, ένα τελευταίο στοιχείο, από πλευρά τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία ε, υποστηρίζουμε ιδιαίτερα την πρόταση του κυρίου Μποβέ, προκειμένου η γνωμοδότηση να προτείνει την εφαρμογή στην περιοχή της Νοτίου Μεσογείου μέτρων ε, ανάπτυξης της Υπέθρου, όπως το Λίντερ. Ο Επίτροπος Τσόλος και εγώ πέρσι ξεκινήσαμε μία διαδικασία EMPART για την ακροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη στην υπαίθρο, με την ανάπτυξη επίσης ε, δυναμικού σε ό,τι αφορά τις γειτονικέ χώρες προς Ανατολάς και προς τον Νότο, σε ό,τι αφορά βάση μάλλον των ε, προενταξιακών μέτρων που χρησιμοποιούνται για τις χώρες υποένταξη. Τα προγράμματα αυτά λειτουργήσαν στην Νότια Μεσόγειο, άρα θα θέλαμε να αναφερθεί συγκεκριμένα, αν θέλετε, το πρόγραμμα LEADER, γιατί το προωθούν οι ίδιοι οι αγρότες. Με αυτά τα σχόλια λοιπόν, Πρόεδρε, σε αυτά τα σχόλια θα σταματήσω και θα περιοριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Εισηγητά, κύριε Δανέλη, θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ την Επιτροπή και τους ε, καλούς συναδέλφους για την ε, συμφωνία στη γνωμοδότηση. Νομίζω ότι είναι ζητήματα, στα οποία δεν μπορεί παρά να έχουμε την ενιαία αντίληψη που μας διακρίνει. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να ξεπεράσουμε και μεγάλες προκλήσεις εξαιτίας και της απουσίας θεσμών αλλά και της ε, ελλειπούς ε, ε, δημοκρατικής κουλτούρας που διακρίνει την περιοχή. Για μας είναι κορυφαίο ζήτημα το να υπάρξει η δυνατότητα της διάχυσης, της ενίσχυσης και η πρόσβαση των μικρομεσαίων καλλιεργητών ή εκείνων που έχουν περισσότερη ανάγκη της στήριξης να μπορέσουν να την προσεγγίσουν. Βεβαίως συμφωνούμε απόλυτα ότι για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια μεγάλη πρόκληση να οργανωθεί μια περιφέρεια ουσιαστικά αγορών στη Βόρεια Αφρική, με την οποία ε, θα έχει σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, βεβαίως η, η υδάτινη πόρη, η ενέργεια, η συνολικότερα η φυσική πόρη είναι ένα, μια βασική, ένα βασικό ζητούμενο από μας το πώς ορθολογικά θα αξιοποιηθούν και θα αναπτυχθούν. Ε, και βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του συναδέλφου Μποβέ. Το Λίντερ είναι μια πολύ θετική εμπειρία ε, για την ε, περιοχή τη δική μας και η τεχνογνωσία που ήδη έχουμε, τα συμπεράσματα που μπορούμε να συνάγουμε, οι καλές πρακτικές μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα, αξιοποιήσιμες στην περίπτωση της στήριξης της νέας αγοράς που δημιουργείται. Ευχαριστώ πολύ. E, Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι καλό θα είναι να σημειώσουμε ότι στα πλαίσια της στρατηγικής επενδύσεων και εμπορίου θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τα θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας, οι εμπειρίες των χωρών που προσχώρησαν στην Ένωση και οι δικές μου εμπειρίες μας καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η μεταφορά τέτοιας τεχνογνωσίας προκειμένου κάποιες λύσεις να καταστούν μόνιμες ως το χαρακτήρα τους. Επίσης, οι διαπροσωπικές επαφές. Είναι σημαντικό να εργαζόμαστε με ανθρώπους, γιατί με άλλες τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να προωθηθεί η δημοκρατία. Και σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, οι συζητήσεις ε, για τη δημοκρατία σε επίπεδο, όταν σε επίπεδο συζητήσεων, δεν επαρκούν. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν την κατεύθυνση των φυσικών πόρων. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, λοιπόν, θα ήθελα να περάσω στο επόμενο θέμα. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ ο εισηγητής μας είναι ο Λούις Άλβες. Θα του ζητήσουμε να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια. Bom dia, colegas. Nós ε, estamos perante um relatório. Καλημέρα, συνάδελφοι. Έχουμε να κάνουμε με μία έκθεση λοιπόν, η οποία για πρώτη φορά αν θέλετε προσπαθεί να συνδέσει το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, για την παγκοσμιοποίηση με τη Γεωργία. Έχουμε ήδη συναντηθεί με το Συμβούλιο και έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν ε, κάποια ερωτηματικά. Το Κοινοβουλίο έχει υιοθετήσει ορισμένα ψηφίσματα σχετικά με διεθνείς υποθέσεις και τη Λατινική Αμερική σαν παράδειγμα και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τις θέσεις μας σχετικά με το ευρωπαϊκό αγροτικό πρότυπο, σεβασμός του περιβάλλοντος, σεβασμός των ελαχίστων κοινωνικών δικαιωμάτων, σεβασμός της ασφάλειας της προμήθειας τροφίμων κτλ. Έχουμε πάρει θέσεις λοιπόν και εμένουμε στις θέσεις αυτές. Και αυτό λοιπόν με οδηγεί στο να σχολιάσω τις προτάσεις τις οποίες κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτάσεις οι οποίες κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση κάποιες ε, από τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπονομεύσουν την διαπραγματευτική ικανότητα του ευρωπαϊκού χώρου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η ανάλυση την οποία μπορούμε να κάνουμε. Ε, ταυτόχρονα διευκολύνοντας αν θέλετε ε, και ε, την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Το Ευρωπαϊκό αυτό Ταμείο καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσει με χρήσιμο τρόπο για τους γεωργούς. Θα πρέπει η πρόσβαση στο Ταμείο να είναι εύκολη και θα πρέπει επίσης να έχει το ταμείο αυτό τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε να βοηθήσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις όταν αυτές είναι απαραίτητες ρυθμίσεις στον τομέα της παραγωγής, του τρόπου παραγωγής ή ακόμα και ε, πλήρης αλλαγή δραστηριότητας όταν ο Γεωργός κρίνει ότι πρέπει να αλλάξει η καλλιέργεια. Εάν θέλουμε λοιπόν το Ταμείο να είναι χρήσιμο, τότε θα πρέπει τα μέσα τα οποία θα καθοριστούν και τα οποία θα είναι στη διάθεσή τους να καθοριστούν και αυτά με πολύ σωστό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν τα μέσα αυτά να είναι αποτελεσματικά και να λειτουργούν σωστά έτσι ώστε να προσφέρουν τις απαιτούμενες λύσεις. Εφόσον θέλουμε το Ταμείο αυτό να λειτουργήσει με τον συγκεκριμένο αυτό ικανοποιητικό τρόπο, και στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών επίσης, θυμίζω ότι αυτό είναι ο στόχος των προτάσεων, θα πρέπει το μέσο αυτό να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την πραγματική κατάσταση. Φυσικά βέβαια πάντα μπορεί να υπάρξουν συμβάντα τα οποία είναι απρόβλεπτα και ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και τα απρόβλεπτα αλλά βασικά θα πρέπει να καλύψει τις προβλεπτές τακτικές αν θέλετε ανάγκες. Εδώ υπάρχουν κάποια σημεία ανησυχίας, ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης. Η διάσταση, αν θέλετε, της απασχόλησης είναι κάτι το οποίο δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη. Στην ουσία ε, στοχεύουμε στις ε, στη μεταφορά των ρυθμίσεων που ισχύουν για τους εργαζομένους στον τομέα της γεωργίας. Αυτό θεωρητικά σωστό είναι. Από την άλλη όμως η απασχόληση στη γεωργία παρουσιάζει κάποια ξεχωριστά θα έλεγα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάτι το οποίο η πρόταση μάλλον δεν αντιμετωπίζει. Ταυτόχρονα θα πρέπει το συγκεκριμένο αυτό ταμείο το οποίο τώρα αν θέλετε ε, θα φτάνει τα δύο δις και τα λοιπά. Έχουμε πει ότι το 80% του ποσού αυτού θα είναι σε θέση να καλύψει ε, τις δραστηριότητες οι οποίες προβλέπονται. Υπάρχουν κάποια ανώτατα όρια σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις οι οποίες θα γίνονται δεκτές Αυτά τα ποσά ακούγονται πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ σημαντικά, αλλά μην ξεχνάτε πως καλύπτουν το σύνολο των γεωργικών δραστηριοτήτων σε 27 χώρες, οπότε δεν είναι τόσο υψηλά. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε έναν σωστό μπούσουλα, αν θέλετε, μπροστά μας, για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα πρέπει να λειτουργήσει το Ταμείο. Το πιο σημαντικό θα έλεγα σημείο του κανονισμού του Ταμείου είναι το 4-3. Αυτό καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας ουσιαστικά του Ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί τη βάση των μελετών τις οποίες έχει ολοκληρώσει μέχρι τώρα, κάνει ένα πρόγραμμα, προτείνει ένα πρόγραμμα μέσω και των κατεξουσιοδότηση πράξεων διευκρινίζει το θέμα των υποψηφιωτήτων και διασφαλίζει έτσι τη σωστή λειτουργία του Ταμείου. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία όπως είπα τα οποία δημιουργούν αμφιβολίες. Έχω την αίσθηση ότι οι αρμοδιότητες τις οποίες θέλει να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον συγκεκριμένο τομέα είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές, περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Είναι πολύ συγκεντρωτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχω κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο να πω σε αυτή τη φάση. Οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν θα κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο αυτό θα επηρεάσει την απασχόληση και θα επηρεάσει το σύνολο του γεωργικού τομέα. Αυτές ήταν κάποιες πρώτες σκέψεις τις οποίες είπα και χρειάζεται να συζητηθούν λεπτομερέστερα σε πολιτικό επίπεδο για να δούμε τι θέλει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρτίνες έχει το λόγο. Όχι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Με κοιτούσατε, αλλά δεν αναγνώρισα το όνομά μου, το ίδιο μου το όνομα. Σας ε, ευχαριστώ. Γκίνες, λέγεται με Γκίνες. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, ότι κινούμαστε εκτός MFF στο ταμείο αυτό. Αυτό με ανησυχεί. Κατά δεύτερον, ότι επεκτείνοντας αυτό το, παγκοσμίο, το, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και, για να συμπεριλάβει και τους αγρότες, πολύ φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα δώσει την ε, προσοχή που αρμόζει στις ε, εμπορικές συμφωνίες και τον αντίκτυπο που θα έχουν στους αγρότες. Ε, δημιουργούμε ένα μηχανισμό πριν από τις συμφωνίες. Αυτό θεωρώ ότι σημαίνει ότι θα είναι επιζήμιες αυτές οι συμφωνίες για τον Ευρωπαίο αγρότη. Θα ήμουν πολύ επιφυλακτική. Δεν θα ήθελα να συμπεριληφθεί αυτή η διάταξη για το λόγω της ανησυχίας αυτής του πώς θα ξεκινήσει και πώς θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το θέμα του Μερκοσούρ, το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι πολύ ανεπαρκές για να καλύψει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο, αρνητικό αντίκτυπο των συμφωνιών αυτών. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων παραγωγών και αγροτών. Πρώτα απ' όλα, αυτό το τονίζω. Το θέμα της χρηματοδότησης είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι και πάλι θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Ας δούμε πόσο περιορισμένη είναι η χρηματοδότηση για την ε, γεωργία, αλλά και το τι θα γίνει και με την χρηματοδότηση άλλων τομέων σε περίπτωση που συμπεριληφθεί η γεωργία. Πραγματικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πολύ πιο λεπτομερείς πληροφορίε από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση αυτή. Πρόκειται για μία ιδέα την οποία λίγοι θα απορρίπταμε, αλλά δεν μπορώ και να την καλοδεχτώ μέχρι να ξέρω πιο πολλές λεπτομέρειες. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται και από εμπορικής πλευράς σε ό,τι αφορά διαπραγματεύσει που θα επηρεάσουν την ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν Χόσλιν. Ναι. Συμφωνώ λίγο πολύ με αυτά που είπε η κυρία Μαγκίνες. Τα αναφέραμε αυτά και με τις συναντήσεις με τον εισηγητή. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να δείξουμε επικριτική στάση σε ό,τι αφορά το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και ότι συμπεριλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή η Γεωργία, αλλά θεωρώ ότι αυτά δεν μπορούμε να τα δεχτούμε έτσι όπως έχουν, σε καμία περίπτωση. Τι μας προτείνετε; Μια κακή συμφωνία, ένα κακό deal. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά επί της αρχής και σε λεπτομέρεια. Το είπα και σήμερα το πρωί στη συνεδρίαση των συντονιστών ότι είναι αυτό θέμα του Προέδρου της Επιτροπής να εξετάσει κατά πόσον στέκει η διαδικασία η οποία εφαρμόζεται επί της αρχής είναι σαφές και αυτό θα πρέπει να το πούμε και στο κοινό ότι ένα πρόγραμμα για τις επιδράσεις ε, της, ε, μάλλον την εξομάλυνση αν θέλετε των επιπτώσεων της απελευθέρωσης της αγοράς και καταρχάς για το Μερκοσούρ υπάρχει μια ανάλυση για το ποιος ε, υπόκειται κάποιες ζημίες μετά από μια συμφωνία Μερκοσούρ. Αλλά αν τα αποδεχόμαστε αυτά, σιωπηρά αποδεχόμαστε και τη συμφωνία Μερκοσούρ. Και νομίζω ότι συμφωνούμε στην Επιτροπή μας ότι είμαστε πολύ επικριτικοί έναντι της συμφωνίας ε, του Μερκοσούρ. Αν δώσουμε λοιπόν ε, ουσιαστικά εντολή αν δώσουμε μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την αρμόδιο Επίτροπο ότι δεν τα δεχόμαστε αυτά χωρίς ε, αντίσταση, νομίζω ότι αυτό θα καταστήσει σαφή και την άποψή μας για τη συμφωνία μας με το Μερκοσούρ σε ό,τι αφορά και τις διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να είναι θετική η εξέλιξη ούτε καν για τον μικρό Γιώργο στην Αμερική. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό, να το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη, γιατί στη μορφή αυτή που μας υποβάλλεται δεν μπορούμε παρά να το απορρίψουμε ως Επιτροπή Γεωργίας. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε λοιπόν αυτό προς τον Επιτροπό Εμπορίου, τον κύριο Ντεχούχτ, ότι δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό. Μια συμφωνία η οποία μακροπρόθεσμα θα μας γλάψει πολύ. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Πέρες Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη συνάδελφο Μαγκίνες. Δεν μπορώ εγώ να συμφωνήσω ότι εδώ πρόκειται για... παρά ότι πρόκειται εδώ για μια δηλητηριασμένη καραμέλα. Απορώ δηλαδή πόσο εισηγητή δεν το είπε. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να εθελοτυφθούμε όταν μας έχουν πειράξει, μας έχουν κάνει κακό και μετά θέλουν να μας δώσουν και ένα χαπάκι δίνοντας ε, τρία δις. Τώρα οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι κερδίζουν τίμια τη ζωή τους ε, με αηφορία που μας επιτρέπουν όλους τους Ευρωπαίους να κρατήσουμε παράδοση και κουλτούρα μέσα από τη δουλειά τους στη Γεωργία και στην ε, κτηνοτροφία και κριτικάρω και την Κομισιόν που θέλει να τελειώνει με αυτές τις συμφωνίες με τους μικροπαραγωγούς στη Νότια Μεσόγειο. Κριτικάρω ε, επίσης ότι θα πρέπει να απογυμνώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους ε, από, την, από το κέρδος του κόπου τους ε, δίνοντάς τους επιδοτήσεις και να τους προτείνουμε εμείς μη γεωργικές δραστηριότητες και όλα αυτά γιατί η Κομισιόν είναι ανίκανη να φανταστεί μια οποιαδήποτε πρωτοτυπία για το πώς μπορεί να προχωρήσει σε μια δίκαιη κατανομή του πλούτου στη Μεσόγειο και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ντροπή να θεωρούμε ότι έχουμε χάσει αυτή την ε, αυτό το παιχνίδι βάζοντας, ε, σκεπάζοντας τα μάτια μας όπως είπε η κυρία Μασγκίνες. Εμείς πρέπει να έχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο για να κινητοποιήσουμε όλα αυτά τα κονδύλια. Πόσες φορές εμείς θα έχουμε την ασφάλεια ότι από 27-28 χώρες συμφωνούν. Τι ευαισθησίες θα έχουν οι χώρες του Βορρά όταν θα έχουμε προβλήματα σε μικρές ε, περιφέρειες ε, του Νότου θα υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Πραγματικά το αμφιβάλλω. Μετά από το θέαμα που είχαμε δηλαδή φέτος το καλοκαίρι με την κρίση του Εκόλη, αμφιβάλλω πάρα πολύ. Και μετά με τη συμφωνία που έγινε του Μαρόκου που υπογράφηκε από τους 27, που υπογράφηκε στο Συμβούλιο από τους 27, αμφιβάλλω κατά πολύ ότι υπάρχουν τέτοιου είδου λεπτότητες και ευαισθησίες. Συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνες και μια που είναι εδώ η Κομισιόλ και μπορούμε να τη ρωτήσουμε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή εμείς ε, θέτουμε εδώ τα κριτήρια επιλεξιμότητας για αυτά τα κονδύλια, λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα ζητούμενα μέχρι, για να δοθούν αυτές οι υποθετικές επιδοτήσεις του υποθετικού ταμείου μέχρι δηλαδή να το βάλει μπρος στο Συμβούλιο. Ο κύριος Μποβέ. Εγώ πιστεύω, όπως και οι τρεις προλαλήσαντες, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μία σαφή θέση για αυτό το ταμείο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η πρόταση είναι πραγματικά μία φόλα των ευρωπαϊκών αρχών προς τους Γιωργούς ε, για να, για να καταπιούνε τις ε, συμφωνίες ελευθέρων ανταλλαγών στις συμφωνίες ανταλλαγών η Γεωργία επιτρέπει στις μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών να κερδίζουν μερίδια της αγοράς και ουέ και λίμωνο για αυτούς τους γεωργούς που χάνονται. Μιλήσαμε για το Μαρόκο, μιλήσαμε για το Μερκοσούρ, αύριο θα μιλάμε για τον Καναδά με το Γάλα και μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τομέα. η γεωργή σήμερα θυσιάζονται στο βωμό των ελευθέρων ανταλλαγών και, ε, του ανοίγματο της αγοράς. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Η Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να αρνηθεί καθαρά και ξάστερα και θα πρέπει να σταθούμε ικανοί σε αυτό το κοινοβούλιο να έχουμε μια πλειοψηφία που να λέει δεν το θέλουμε αυτό το ταμείο. Πρόκειται για ένα δώρο που κάνουμε στις, τρί, στις άλλες χώρες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εμείς ξεκινάμε μια διαπραγμάτευση και η χώρα απέναντι, η Μερκοσούρ για παράδειγμα. Ξέρει ότι υπάρχει ένα κονδύλιο προσαρμογής ε, στη, στη, στη Γεωργία, τότε μπορεί κάλλιστα να κάνει ό,τι θέλει, διότι κανένας δεν πρόκειται εδώ να χτυπηθεί διότι, από το Συμβούλιο, διότι θα πούνε ότι ορίστε, έχουμε ένα ταμείο το οποίο μας επιτρέπει να ξοπετάξουμε τους γιοργούς μας με μία αποζημίωση. Εμείς είμαστε εδώ για να υπογράψουμε την απόλυση των γεωργών από το, το κτήμα τους. Είμαστε εμείς αυτοί που θα σταματήσουμε οποια, οποιαδήποτε μορφή κτηνοτροφίας αυτό το ταμείο συγχρηματοδοτείται από την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τα κράτη θα πρέπει να βάλουν πάλι το χέρι στην τσέπη για να απολύσουν τους γεωργούς τους και αυτοί θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Παίρνω την ε, περίπτωση της Ισπανίας. Αν ψήφιστη στο, κοινοβούλιο η συμφωνία με το Μαρόκο εμείς πρέπει να αποφύγουμε να, να το ψηφίσουμε. Αλλά σήμερα στην Ανδαλουσία έχουμε 40% ανέργους στο γεωργικό τομέα. Θα τους πληρώσουμε με αυτό το ταμείο. με αυτό το ταμείο θα τους επιτρέψουμε να έχουν ένα εισόδημα για κανένα χρόνο. Εγώ νομίζω ότι εδώ πουλιόμαστε σαν γουρούνι στο σακί για σε αυτούς που θέλουν να ανοίξουν την αγορά. Ο εισηγητής έδωσε αρνητική γνώμη και θα πρέπει να κινητοποιηθούμε και θα κινητοποιηθούμε και θα ενημερώσουμε τους γεωργούς για το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι θα πρέπει να καταγγείλουμε ολόψυχα αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο George Λάιον και μετά η κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις απόψεις που παρουσίασαν πολλοί από τους ομιλητές. Πρόκειται για ε, μια πολιτική πλάνη αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί δεν είναι την νομιμότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περικόψει τη χρηματοδότηση. Ίσως κάποιος θα έλεγε ότι δεν έχουν περικοπεί ε, η χρηματοδότηση γιατί προσθέθηκαν τόσο πολλά κονδύλια στην γεωργία. Και κατά δεύτερον δείχνει, δίνει μία λευκή επιταγή στον Επιτροπό ε, στη διαπραγμάτευση των ε, συμφωνιών ότι έχουμε όλες τις λύσεις για τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύψουν και δεν θα πρέπει να ανησυχώ, δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τα, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της διαπραγματευσής μου. Νομίζω ότι ως Επιτροπή Πολιτικής Άποψης, λοιπόν, θα πρέπει να αντιταχθούμε στην ε, συνολική πρόταση. Αλλά παρουσιάζεται ένα σημαντικό πρόβλημα. Πώς θα το κάνουμε αυτό, γιατί η πρόταση αυτή δεν, είναι, δεν είμαστε αρμόδια εμείς. Έχουμε συζητήσει και με την ε, Επιτροπή Απασχόλησης και με την αρμόδια ε, Επιτροπή. Θα δώσουμε κάποιες αρμοδιότητες για κάποια άρθρα, για το Ξέρουμε ότι έχουν αυτά αποσυρθεί. Να συζητήσουμε λοιπόν στη διάσκεψη των Προεδρών για να δούμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε την Επιτροπή Απασχόλησης. Νομίζω ότι κάποια στιγμή το Μάιο, τον Ιούνιο έχει προβλεφθεί. Ένα τμήμα λοιπόν της ε, μεταρρύθμισης της ΚΑΠ θα έχει ήδη τύχη διαπραγμάτευσης προτού αρχίσουμε να κάνουμε τέτοιες αλλαγές. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν ε, μηχανισμοί για το CEP και θα θέλαμε να εξετάσουμε ενδεχόμενο αντίκτυπο των μελλοντικών συμφωνιών. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Υπάρχει το επιχείρημα ότι τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά είναι εκτός του προπολογισμού για τη γεωργία. Αυτό θα μπορούσε να μας καθυστερήσει, αλλά θεωρητικά πιστεύω, στην πραγματικότητα μάλλον πιστεύω, ότι αυτή η γραμμή του προπολογισμού είναι πραγματικά παραπλανητική. Δεν νομίζω ότι θα υποφεληθεί ιδιαίτερα ο τομέας ε, της γεωργίας από την ε, γραμμή αυτή του προϋπολογισμού. Γι' αυτό, αυτή θεωρώ ότι είναι σκληρή πραγματικότητα Ρωτάω και ζητάω λοιπόν από την Γραμματεία να μας επιβεβαιώσει τι δυνατότητες έχουμε ως Επιτροπή δεδομένων των δύσκολων συνθήκων επειδή δεν έχουμε την αρμοδιότητα εκτός και αν το περάσουμε αυτό από τη διάσκεψη των Προέδρων για να ζητήσουμε εκ νέου τον έλεγχο των συγκεκριμένων τμήματων της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την Επιτροπή μα, Αν δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε και να ζητήσουμε τον έλεγχο και την αρμοδιότητα, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στην Ολομέλεια. Και εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα, θεωρώ. Ζητώ λοιπόν από τον Πρόεδρο και από την ομάδα του να υποβάλουν κάποιε πρακτικέ προτάσει για το πώ θα πραγματοποιήσουμε και θα εφαρμόσουμε όλες τις απόψεις που ακούσαμε. Ιδάλλως είναι θεωρητικό το εγχείρημα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ουσιαστικά. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να μπει στην, τον κανονισμό για την ΚΑΠ κάποια αρετή αναφορά προκειμένου οι μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε να τη χάνουν διαπραγμάτευση και αντιμετώπιση με τα υφιστάμενα μέτρα. Και πάλι θέλω και ζητώ την βοήθεια και τις συμβουλές από πλευράς του Προέδρου και από τη Γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ. Πατρανέβες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εάν θα έπρεπε να προσπαθήσω να αποδώσω περιληπτικά θα έλεγα την αίσθηση που έχω για το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλά συγκεκριμένα πράγματα μπροστά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάποιες παρουσιάσεις ε, οι οποίες ε, είναι σε επίπεδο ιδεών. Λένε τι ωραία θα ήταν να είχαμε ένα ταμείο, να έχουμε κάποια χρήματα στη διάθεσή μας, κάτι το οποίο θα ήταν θετικό για τη Γεωργία. Ε, να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι το σοβαρό. Δεν υπάρχει τίποτα για μας εδώ. Από το 2007 υπάρχει αυτό το ταμείο. Το ταμείο περιορίζει την δραστηριότητά του στον τομέα της απασχόλησης. Στην ουσία λένε ότι εδώ θα καλυφθούν κάποιες συνέπειες στην ΚΑΠ από διεθνείς συμφωνίες. Από την άλλη προκαταλαμβάνουμε αν θέλετε ότι οι αρνητικές συνέπειες των διεθνών συμφωνιών και στον τομέα της γεωργίας είναι κάτι το αναπόφευκτο. τα χρήματα τα οποία είναι στη διάθεση δεν είναι ε, πάρα πολύ υψηλά. Το επίπεδο συγχρηματοδότησης από την εθνική πλευρά είναι πάρα πολύ υψηλό. Οπότε έχουμε να κάνουμε τώρα με μία πρόταση η οποία θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Γιατί κανένας δεν ξέρει ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο μέσο. Κανένας δεν ξέρει το μέσο αυτό αν θα είναι σε θέση να καταστεί λειτουργικό. Και η γεωργία στην ουσία χρησιμοποιείται για μια ακόμη φορά σαν ανταλλακτικό μέσο θα έλεγα και ακούγονται διάφορα παρηγορητικά λόγια για τη γεωργία όταν οι διεθνείς συμφωνίες λειτουργούν εις βάρος της. Πάρτε το παράδειγμα της συμφωνίας με το Μαρόκο. Υπάρχει το παράδειγμα της συμφωνίας με το Μερκοσούρ. Τα συμφωνίες αυτές ε, θα δημιουργήσουν προβλήματα στη Γεωργία και γι' αυτό έχουμε το συγκεκριμένο ταμείο. Τίποτα δεν θα κάνει το ταμείο. Μιλάμε για μία σαχλαμάρα, μιλάμε για μία απάτη. Πρέπει να αντιδράσουμε στις προτάσεις αυτές γιατί είναι προτάσεις κενές περιεχομένου κύριος Λάιονς μας είπε ότι υπάρχουν ε, και προβλήματα συντονισμού με την Επιτροπή Απασχόλησης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ίσως να έχει δίκιο. Αυτό όμως το οποίο εγώ διαπιστώνω είναι ότι το μέσο αυτό υπάρχει έτσι και αλλιώς στον τομέα της απασχόλησης εδώ και αρκετά χρόνια και θα πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται με τους στόχους με τους οποίους ε, ε, ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια. Το να διευρυνθεί στη γεωργία δεν βοηθάει σε τίποτα και κυρίως δεν βοηθάει τους ίδιους τους γεωργούς. Μιλάμε για ταμείο προσαρμογής στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Όχι. Το μόνο που κάνει είναι να αντιμετωπίζει κάποιες από τις συνέπειες των διεθνών συμφωνιών. Αυτό είναι όλο, τίποτα περισσότερο. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση αυτή. Θα πρέπει να διατυπώσουμε εμείς εδώ μια διαφορετική στρατηγική, πολύ πιο συγκεκριμένη. Έχουμε κάποιες αρνητικές, αν θέλετε, συνέπειες σε σχέση με τη γεωργία των διεθνών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό είναι το θέμα το οποίο θα πρέπει να αναλύσουμε. Ας μην παρασυρθούμε λοιπόν από τις κενές περιεχομένου ιδέες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ας μην την αφήσουμε να βγαίνει αθώα από αυτά τα οποία έχει κάνει μέχρι τώρα. Επιτρέψτε μου να λειτουργήσω και λίγο θετικά, με επικοδομητικό πνεύμα. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εν μέρη θετική, διότι είναι, θα έλεγα, υποδειγματική κατά κάποιο τρόπο. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο Επίτροπος Ντεγκούχτ την Γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα σημαντικό κείμενο που είχε δημοσιευθεί στις 12 Δεκεμβρίου, Οκτωβρίου, συγγνώμη, ρύθμιση της ΚΑΠ, έλεγε ότι η αγροτική πολιτική πρώτον έχει σαν στόχο να θρέφει 450 εκατομμύρια πολίτες, ίσως να συμπληρώνουμε με κάποιες εμπασπεριτώσεις συμπληρωματικές εισαγωγές. Μας θυμίζει επίσης ότι είμαστε μια παλαιά ήπειρος και ανταποκρίνεται επίσης και σε ένα εδαφικό στόχο. Την παρουσία στην Ήπεθρο δηλαδή ε, των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μας θυμίζει επίσης ότι η γεωργία και η επεξεργασία γεωργικών προϊόντων είναι η πρώτη πηγή θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πρέπει να θέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προευθυνών της και δεν ασχολήθηκα, θυμίζω, και με, την, με το θέμα του περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να λέει από τη μία στην ουσία τρεις βασικούς στόχους και από την άλλη να θέτει ένα συμπληρωματικό στόχο μετακόμισης, αν θέλετε, της Υπέθρο. Όχι, η ύπεθρος δεν μεταφέρεται. Στα πλαίσια της λογικής που λέγουμε εδώ και δυόμιση χρόνια και μετά από την έκθεση για το Μαρόκο δεν μπορούμε παρά να αρνηθούμε en bloc συνολικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ με δύο καπέλα, σαν εισηγήτρια στην Επιτροπή Απασχόλησης και σαν αναπληρώτρια μέλος της Επιτροπής Γεωργίας. Όταν ασχολήθηκα με το θέμα αυτό μετά την ανακοίνωση του Επιτρόπου, αμέσως σηκώθηκε αν θέλετε, άναψε ένα κόκκινο φωτάκι σε σχέση με τη Γεωργία. Άκουσα κάποια από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεται. Θα συμφωνήσω με την συνάδελφο Πατραονέβες ότι αυτό το οποίο σας προτείνουν είναι ένα δηλητηριασμένο δώρο. Αυτό το οποίο σας προτείνουν είναι ένα φύλλο σικής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να συνεχίσει με τις διαπραγματεύσεις της χωρίς προβλήματα και να πει και στο Κοινοβούλιο και τους Γεωργούς ότι κοιτάξτε εμείς σας δίνουμε στην διάθεσή σας το Ταμείο το οποίο θα επιτρέψει να ε, επανεκπαιδευτείτε αν χάσετε την δραστηριότητά σας. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ παρά να αρνηθώ. Θα ήθελα να πω επίσης ότι βλέποντας και την αξιολόγηση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας διαπιστώνω ότι κάποιες από τις περιοχές οι οποίες θα φυγούν είναι αυτές οι οποίες είναι πάντα στα πλαίσια της συνοχής. Ξέρετε ότι ένα σκέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λειτουργεί στα πλαίσια της συνοχής και ένα άλλο σκέλος θα συνάπτει εμπορικές συμφωνίες που θα βλάπτουν τις περιοχές της συνοχής. Λοιπόν, και τώρα εμπλέκεται και το Κοινοβούλιο. Είχα αρκετές συναντήσεις με τον κύριο Άλβες συζητήσαμε τις δυνατότητες να προσπαθήσουμε να μοιράσουμε κάπως την έκθεση αυτή. Παρ' όλα αυτά η θέση της Επιτροπής Απασχόλησης μετά από την συνάντηση των συντονιστών είναι ότι η απασχόληση θα ζητήσει την πλήρη αρμοδιότητα. Οι συζητήσεις που είχαμε τους κοιόδης εισηγητές δείχνουν ότι δεν θέλουν να εξαιρέσουν τους γεωργούς, αν και κάποιοι σκιώδεις είχαν πολλές επιφυλάξεις για τον ρόλο της Γεωργίας εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει εφόσον συμπεριληφθούν οι Γεωργοί θα συμπεριληφθούν με τις ίδιες προϋποθέσεις με τους εργαζόμενους γενικότερα εκτός Γεωργίας. Κάτι το οποίο δεν έχει νόημα βέβαια γιατί όταν κάποιος σταματήσει να εργάζεται στη Γεωργία είναι δύσκολο να επανέλθει. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξει κανείς σε μια κάποια διαδικασία. Όταν λύσουμε το θέμα της αρμοδιότητας ίσως να διευκολυθούν κάπως οι τρόποι με τους οποίους θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κύριος Νίκολσον. Να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρο. Πολλά από αυτά που σκόπευα να πω τα ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Χάρκιν. Αυτό ασφαλώς αφορά την ε, πλευρά του κλάφου της γεωργίας, της ε, βιομηχανίας. Και αποτελεί και μια συνταγή, αν θέλετε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βγει και να κάνει διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ε, σε όλο τον κόσμο που θα θεωρεί ότι είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς και η πρώτη θα είναι η Μερκοσούρ, θα είναι η τελευταία όμως. Υπάρχει ένα θέμα αρχής, ξέρετε, εδώ πέρα. Και δεν έχει να κάνει με το πού ξεκινά και πού τελειώνει η αρμοδιότητα του καθενός και πώς διαιρείται. Το Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση σκοπό είχε να αν σκοπό είχε να βοηθήσει τους αγρότες, το οποίο αμφιβάλλω ειλικρινά, γιατί δεν βλέπω πώς θα έχει πρόσβαση ο Γεωργός σε αυτό, αν ε, ε εξισώνεται με τον ε, εργάτη στα εργοστάσια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα λειτουργήσει στο δικό μου κράτος μέλος κάτι τέτοιο. Στην Ευρωπαϊκή, μάλλον η Επιτροπή μας θα γελιοποιηθεί αν μας πούνε ότι υπάρχει ένα ταμείο παγκοσμιοποίηση για τους γεωργούς και το αποδεχτούμε και σε τελική ανάλυση δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν κονδύλια πραγματικά. Κονδύλια στα οποία να υπάρχει πρόσβαση αν χρειαστεί. Άρα ανησυχώ, ανησυχώ ιδιαίτερα. Και υποστηρίζω και τον εισηγητή και την κυρία Χάρκιν γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε επί της αρχής εδώ στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι πρόκειται για μια ανησυχία η οποία άλλο ένα και υποδαβλίζεται εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι θα πρέπει η αρμοδιότητα σε υψηλό επίπεδο να μοιράζεται μεταξύ των επιτροπών. Αυτό το πράγμα που μία επιτροπή αρπάζει όλη την αρμοδιότητα παράλληλα που δεν είναι όλα τα θέματα στο δικό της ε, πεδίο θέτει πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας ε, του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος και πολλές φορές έχουμε τσακωθεί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τώρα αναπάντεχα έτσι εξελίσσεται και η κατάσταση με την Επιτροπή Απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασιστούν αυτά σε υψηλό επίπεδο και αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων θα πρέπει να αξιολογήσουν πλήρως με βάση τα στοιχεία την κατάσταση. Είναι λοιπόν ένα σημείο καμπής. Θα πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν υπό το πρίσμα αυτό και να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πουτσίσκη. Από την Γεωργίας. ο εκπρόσωπος της Κομοσιόν, όχι... Σας ευχαριστώ και πολύ λυπάμαι που ήρθα καθυστερημένα. Εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, η οποία είναι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση για το Ταμείο ως τώρα. Σε στενή συνεργασία με, την, με τους συνοδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, οι οποίοι ο, επίσης παρίστανται. Να κοιτάξουμε λίγο πώς ε, δημιουργήθηκε το Ταμείο και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε και τι έχει πετύχει ως τώρα. Και θα ζητήσω μετά από τους συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν σε ό,τι αφορά τις γεωργικές πτυχές των νέων προτάσεων. Το Ταμείο δημιουργήθηκε στις αρχές του 2007, τέθηκε σε εφαρμογή ως απάντηση στις εμπορικές συμφωνίες, τα εμπορικά προβλήματα, σε προβλήματα που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση, από εμπορικά ζητήματα και στην αρχή το τομείο μπορούσε να ανταποκριθεί σε αιτήσει χιλιάδων υπαλλήλων, εργατών, χίλιων μάλλον ε, ε, υπαλλήλων εργατών μετά περιορίστηκε σε 500 υπαλλήλου σε περίοδο 9 ή 12 μηνών. Τα μέτρα είναι ενεργά μέτρα πολιτικής. Δεν μπορούν να ζητούν μεμονωμένοι όμως εργάτες να υποβάλουν αίτηση. Το κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση και οργανώνει τα μέτρα για τους εργάτες. Το κράτος μέλος έχει κοινή ευθύνη μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο βαθμός συγχρηματοδότησης είναι στο 50% σήμερα. Ήταν 65% για μία περίοδο όπου υπήρχε η απόκληση λόγω κρίσης. Λόγω της παγκόσμιας κρίσης μπορέσαμε να δώσουμε συγχρηματοδότηση ύψους 65%. Δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο για να παρατεθεί αυτό μέχρι τα τέλη του 2013, άρα έχουμε επανέλθει σε συγχρηματοδότηση 50%. Τα χρόνια λοιπόν αυτά είχαμε 97, λάβαμε 97 αιτήσει από 20 κρατημέλη. 90.000 εργάτες ε, και 450 εκατομμύρια έχουμε δαπανίσει 83 εκατομμύρια ανά 17% δηλαδή του maximum για τη θέμενου ποσού, το οποίο πάντα ήταν κατά προσέγγιση αρκετά υψηλό προκειμένου να μπορέσει να καλύψει ενδεχόμενες κρίσεις, ενδεχόμενα απρόβλεπτα περιστατικά, γιατί ασφαλώς το Ταμείο ε, προορίζεται για τέτοια απρόβλεπτα περιστατικά έγινε μία ενδιάμεση αναθεώρηση προσφάτως. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής ήταν τα εξής. Το Ταμείο ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά σε μεγάλες κλίμακας απολύσεις, βοηθώντας ιδιαίτερα τις υπηρεσίες απασχόλησης στα κράτη-μέλη, οι οποίες θα είχαν ε, υποστεί υπερβολικά μεγάλο φόρτο λόγω των μεγάλων των ευρέων αποκλήσεων. Η βοήθεια λοιπόν ήταν σημαντική. Ήταν πολύ πιο προσωπική στη φύση της, πιο μακροπρόθεσμη. Σε κάποιες περιπτώσεις τα μέτρα ήταν καινούργια και παρατάθηκαν. Οι κοινωνικοί εταίροι ενεπλάκησαν και αυτό έκανε τα μέτρα πιο ποιοτικά και ήταν άρα και πιο μεγάλη η αποδοχή. Υπήρξε αλληλεγγύη από πλευράς Ένωσης προς τα κράτη-μέλη και προς τους εργάτες, αλλά επειδή πρόκειται για κονδύλια ανακύκλωσης εκτός των πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών, υπήρξε αλληλεγγύη και μεταξύ των κρατών μελών. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πτυχή της επικουρικότητας ελήφθη υπόψη είναι επαρκώς, γιατί τα κράτη-μέλη είναι αυτά που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τα μέτρα, άρα δεν τους έχει επιβληθεί το οτιδήποτε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα για το νέο πακέτο από το 2014 μας ζητήθηκε να υπάρξει επέκταση και στον τομέα της γεωργίας γιατί κατά το παρελθόν δεν υπήρχε δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από πλευρά τους των αγροτών γιατί οι αυτοαπασχολούμενοι δεν περιλαμβάνονταν πλέον περιλαμβάνονται όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι διαχειριστέ μικρών επιχειρήσεων. Συμπεριλαμβάνονται λοιπόν και οι γεωργοί. Το Ταμείο εξακολουθεί να παραμένει εκτός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού γιατί τα κονδύλια τα οποία δαπανώνται δεν μπορούν να προβλεφθούν. Δεν ξέρουμε πότε θα χτυπήσει η κρίση, πότε θα γίνουν μαζικές απολύσεις. Ακόμα και για τις εμπορικές συμφωνίες δεν ξέρουμε πότε θα προκύψουν. Άρα δεν έχει νόημα να υπάρχει ένα σταθερό προπολογισμό για κάθε χρόνο όταν ένα έτο ενδεχομένω να μην αρκούσε αυτό ο προπολογισμό και κάποιο άλλο έτο ενδεχομένω και να παρήσευε. Μένουμε λοιπόν εκτό των ε, πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών με maximum 3 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2014 μέχρι το 2020. 2,5 δισεκατομμύρια maximum θα μπορέσουν να δαπανηθούν από το ποσό αυτό στους γεωργούς. Τι θα παραμείνει απαράλλαχτο στο μέλλον τα κράτη-μέλη θα εξακολουθήσουν να υποβάλουν αιτήσει και όχι οι εταιρείε ούτε οι ιδιώτες. Η περίοδος αναφοράς θα, θα παραμείνει 4 έως 9 μήνες. Για τον τομέα εκτός της γεωργίας θα, ξαναμείνει... θα ε, εξακολουθήσει να υπάρχει το όριο των 200.000 απολύσεων και ισχύει ότι ενδεχομένως ε, λόγω ειδικών συνθήκων να μην ισχύσουν τα σημεία αυτά, αυτά τα κατόφλια. Βαθμός εκμεταβότησης, μάξιμου 65% θα υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον δε για μία ρήτρα για τις κρίσεις. Ε, μπορεί να μην πρόκειται για μία συγκεκριμένη κρίση όπως αυτή που διανύουμε στην τρέχουσα περίοδο, μια οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση, μπορεί να είναι μια περιφερειακή, μια τοπική κρίση, μια περιβαλλοντική κρίση, όπου το Ταμείο Αλληλεγγύης θα μπορέσει να παρέμβει για εμπορεύματα, αγαθά, για περιουσίες που καταστρέφονται, αλλά που δεν μπορεί να παρέμβει για απολύσεις μαζικές εργαζομένων. Τα μέτρα θα εξακολουθήσουν να είναι ενεργά μέτρα εργατικής πολιτικής, δεν θα υπάρξουν καθαρές παροχές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέτρα για την εξέβρεση νέες θέσεις απασχόλησης ή για τη λήψη μέτρων που θα βοηθήσουν να ανταποκριθεί καλύτερα στο διεθνή ανταγωνισμό. Θα υπάρχουν κάποιες τεχνικές προδιαγραφέ για την επίσπευση και την απλούστευση τη διαδικασίας και για την ευελιξία της ε, διαδικασίας. Θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των κονδυλίων σε πιο επιτυχή, αν θέλετε, μέτρα. Επίσης, προβλέπουμε και μία ενδιάμεση έκθεση προκειμένου και στο μέλλον να είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε καλύτερα το τι θα συμβεί τους 24 μήνες εφαρμογής των μέτρων. Αυτά λοιπόν εν γέννη, αυτές είναι οι δυνατότητες του Ταμείου και για το μέλλον και θα ήθελα να δώσουμε το λόγο, Πρόεδρε, να μου επιτρέπετε και στους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τις πιο συγκεκριμένες πτυχές. Σας ευχαριστώ και πολύ λυπάμαι που έκανα λάθος το όνομά σας. Από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Thank you, Chair. Good morning, ladies and gentlemen. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Προέρχομαι από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας λοιπόν. Σας ευχαριστώ για τις ειλικρινείς ε, αντιδράσεις και σχόλιά σας μέχρι τώρα. Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο γιατί θέλουμε να συμπεριλάβουμε τους γεωργούς στο ταμείο αυτό. Το θέμα είναι ότι ε, υπήρχε εξαίρεση μέχρι τώρα για τους γεωργούς και αυτός είναι ένας λόγος αν θέλετε για να συμπεριληφθούν στο μέλλον. Υπάρχουν αρκετές συμφωνίες, οι οποίες είναι σε διαδικασία υπογραφής τώρα, που εξηγούν την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι γεωργοί στο μέλλον. Αυτά περιλαμβάνονται και στην πρόταση την οποία έκανε τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λέγεται ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζομένων όταν θίγεται η ζωή τους από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Έχουμε, θα έλεγα, αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στους εργαζομένους στη Γεωργία και εκτός Γεωργίας, αλλά και αρκετές διαφορές βέβαια. Το θέμα είναι όμως ότι παρά τις διαφορές η πηγή του προβλήματος είναι η ίδια, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση. Μιλάμε για λύσεις τις οποίες προτείνουμε παρόμοιες ανατομέα, μιλάμε δηλαδή για την εκπαίδευση, για την κατάρτιση, έτσι κι αλλιώ είναι ένα ταμείο θα έλεγα κατεπήγων ω εκ τούτου η διάρκεια του θα είναι πολύ συγκεκριμένη τα ποσά επίσης είναι συγκεκριμένα δεν μιλάμε για αντισταθμίσεις για μια εμπορική, σε μια εμπορική συμφωνία μιλάμε για συγκεκριμένα ποσά και αν θέλετε η λογική πίσω από την εισαγωγή των γεωργών είναι μια στοχευμένη υποστήριξη προς τους γεωργούς έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς. Είναι ένα επιπλέον μέσο δηλαδή για τους γεωργούς να προσαρμοστούν στην αγορά. Πολλές φορές οι γεωργοί είναι αυτοαπασχολούμενοι, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ο τομέας είναι επίσης πάρα πολύ, δια, πολύ διασπασμένος θα έλεγα, οπότε υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Και αυτός είναι ο λόγος, εν πάση περιπτώσει, για τον οποίο θεωρήσαμε ότι στα πλαίσια του γεωργικού τομέα θα πρέπει να ενταχθεί στον, στη λειτουργία του Ταμείου. Έχουν υπάρξει και διαφορετικές απόψεις και από το Κοινοβούλιο και από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υπάρχουν αντιδράσεις, φοβούνται ότι η Γεωργία θα πάρει θα λέγαμε τα περισσότερα χρήματα, το μεγαλύτερο ποσοστό. Θεωρούν ότι είναι ένα δώρο επιπλέον προς τους Γεωργούς Οι εμπορικές συμφωνίες ε, ε, έτσι και αλλιώς ε, όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος τόσο περισσότερο θα ποσοτικοποιούνται επαρκώς και γι' αυτό θέλουμε να προκαταλάβουμε τις αντιδράσεις μας. Δεν θέλουμε εμείς να αντιδρούμε εκ των υστέρων. Εδώ δεν θα πρέπει να περιμένουμε να χάσουν τη δουλειά τους οι γεωργοί. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προκαταλάβουμε κάπως τις καταστάσεις έτσι ώστε και οι γεωργοί να είναι έτοιμοι όταν υπάρξουν κάποιες σοβαρές αλλαγές στην καθημερινότητά τους και στη δουλειά τους. Τώρα για την καταμέτρηση, αν θέλετε, των επιπτώσεων σε επίπεδο ποσοτικό. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες μέχρι τώρα. Αναφερθήκατε στην περίπτωση του Μερκοσούρ. εμεί στη Γενική Διεύθυνση γεωργία αλλά και στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου έχουμε κάνει αρκετέ μελέτες τι οποίες έχουμε καταστήσει διαθέσιμε προς το Κοινοβούλιο από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και στη δική σας Επιτροπή και στην Ίντα. Θεωρούμε ότι τα θέματα τα οποία περιλαμβάνουμε εκεί είναι σημαντικά και θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία προς ενημέρωσή σας και θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε σε σχέση με όλες αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε περαιτέρω ε, ε, ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τους διερμηνείς να μείνουν λίγα λεπτά παραπάνω. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι ανήκω στη λεγεών εκείνων που προσπάθησαν να συντονίσουν τα πράγματα με όλους τους ενδιαφερόμενους για το Μερκοσούρ για παράδειγμα όπου υπήρξε και ένα ψήφισμα για να ξαναδούμε τις παραχωρήσεις εκείνης της συμφωνίας και να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους γεωργούς. Γνωρίζουμε λοιπόν καλά ποιες είναι οι θέσεις, το τι παίζεται. Εμείς πρέπει να υπερασπίσουμε τις συμφωνίες, σύμφωνοι αλλά αυτή η έκθεση δεν είναι μια έκθεση δικής μου πρωτοβουλίας. Η πρόταση δεν, γίνεται, δεν, δεν διατυπώνεται από μένα. Πρόκειται για μια έκθεση μέσω της οποίας εγώ θέλω να δώσω τους καλύτερους όρους ε, για τους ε, δικούς μας ε, γεωργούς. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη κατάσταση. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τους όρους της συζήτησης, ούτως ώστε να εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, έγιναν συνεδριάσεις το Νοέμβριο, προβλέπονται συνεδριάσεις το Μάρτιο, υπάρχουν περιφέρειες που και σήμερα απειλούνται από μεγάλη μείωση εισοδήματος. Σε αυτή λοιπόν την αξιολόγηση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία. όλα αυτά για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που έχουμε μπροστά μας. Εμείς δεν είχαμε βέβαια επαφές με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εμείς ε, δεν μπορούμε να μείνουμε εκτός συζήτηση. Θα έλεγα λοιπόν ότι πέρα από τα εισαγωγικά θα έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε επί του συγκεκριμένου για να δώσουμε τις πιο χρήσιμες λύσεις ε, για τους γεωργούς. Θα πρέπει να δούμε αν είναι χρήσιμο αυτοί οι γεωργοί να εμπλέκονται άμεσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μήπως θα έπρεπε να βρούμε μία δράση σε επίπεδο ΚΑΠ. Χρειάζεται μία δική μας ισχυρή θέση, όχι διασπασμένη θέση. Ευχαριστώ, ψάχνω λοιπόν διευρυμένη συνένεση. Ευχαριστώ πολύ. Όπως θα διαπιστώσατε από τη συζήτηση, το θέμα χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά και προσαρμογές στον τομέα της γεωργίας. Ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ, θα τα ξαναπούμε στις 3 και θα έρθει η Δανή υπουργό. η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου Γεωργίας. Ευχαριστώ τους Διερμήνης.